Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ορίσατε ε, στην επόμενη συνεδρίαση ε, ε, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, έκτακτη συνεδρίαση. Δυστυχώς ο πρόεδρος κολλείεται και γι' αυτό τον αντικαθιστώ εγώ. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, συμφωνείτε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ωραία. Το γλωσσικό προφίλ της συνεδρίασης. Δεν έχουμε διερμηνία προς τα κροατικά, δανικά, λιθουανικά, λετονικά, μαλτεζικά, σλοβακικά και εγωιδελικά δυστυχώς. Και ε, θα περάσω αμέσως στο πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται μία ώρα συζήτησης για αυτό το θέμα, για τη νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το σύστημα προφοριών και άδεια ταξιδίου, αιτίας λέγεται αυτό. Είμαι η συγκήτρια. Η πρόταση κατατέθηκε στην Επιτροπή μας στις 22 Μαρτίου. Αν μου επιτρέπετε θα σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σίμονς που είναι ο εισηγητής από την ΟΚΕ να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση της γνωμοδότησης Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Την ΟΚΕ δηλαδή, ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Και στο τέλος θα ζητήσω από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις τους η συζήτηση με τους συνάδελφους. Καλώς ορίστε κύριε Ντεπρέ, σκιώδης συζητής. Ξέρω ότι η κυρία Γκυγιόμ και η κυρία Βερζιά κολλίονται και ζήτησαν συγγνώμη, δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Η κυρία Ζήπελ αντικαθιστά την κυρία Γκυγιόμ. Ωραία. Να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου. Με λίγα λόγια, Έχουμε ένα σημαντικό θέμα μπροστά μας και έχει σημασία λόγω της περιπλοκότητας να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μέσω συζήτησης. Έτσι πιστεύω. Ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ θεμητός και καλός στόχος να υπάρξει ένα σύστημα ευρωπαϊκό ενημέρωσης για τα ταξίδια, τις μετακινήσεις. Η πρόταση της Επιτροπής κατετέθη το Νοέμβριο και βασικός στόχος είναι κάτι το οποίο δεχόμαστε. Μας δίνει τη δυνατότητα το έτιας να αξιολογήσουμε τις εξαιρέσεις της στο σύστημα θεωρήσεων των πολιτών τρίτων χωρών που θέλουν να έρθουν στη ζώνη Σέγγεν και είναι ένα μέσο ελέγχου αν θέλετε των κινδύνων για πιθανή παράνομη ή παράτυπη μάλλον μεταφορά και μετανάστευση πριν φτάσει στα σύνορα το συγκεκριμένο πρόσωπο, ελέγχονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αιτείται την χορήγηση θεώρησης. Αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα είναι ότι οι συνοριοφύλακες καλούνται επιτόπου μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν πολλαπλού τύπου αξιολογήσεις και εκτιμήσεις. Το σύστημα αίτιας θα δώσει την δυνατότητα να γίνονται κάποιοι προκαταρκτικοί έλεγχοι, οι οποίοι αλλιώς δεν θα ήταν εφικτό να γίνουν. Θα δίδονται ε, πληροφορίες ε, στον συνοριοφύλακα Βέβαια το σύστημα δεν θα εμποδίζει ε, το συγκεκριμένο σύνοριοφύλακα να παίρνει την τελική απόφαση εφόσον εκτιμά ότι ε, δεν υπάρχουν προβλήματα στη συνέχιση της διαδικασίας εισόδου. Το σύστημα νομίζουμε ότι θα μειώσει το ποσοστό ε, των αρνήσεων χορήγησης γιατί θα γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο πριν ξεκινήσει για να διασχίσει τα σύνορα Σέγγεν. Αυτό θα βελτιώσει γενικά λοιπόν την διαχείριση των σύνορων και γι' αυτό υποστηρίζω την βασική λογική και τους βασικούς στόχους της Επιτροπής. Προτείνω και μία σειρά τροπολογιών για περαιτέρω βελτίωση θα πρέπει να πούμε ότι η έκθεση αυτή καθεαυτή σε αυτή τη φάση έχει ε, χώρους βελτίωσης, διευκρινήσεων και για να προετοιμάσουμε λοιπόν αυτή την πρόταση έκθεσης πήρα πληροφορίες από πολλές πηγές, είχα πολλές συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο με τις υπηρεσίες της Επιτροπής έγιναν συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι συζητήσεις μαζί τους ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Πριν φτάσουμε στην παρούσα φάση. Είχαμε συναντήσεις επίσης και με τις εξωτερικές υπηρεσίες που ενδιαφέρονται για το ΕΤΙΑΣ, όπως τη Eurojust, τη Europol, Είχαμε επίσης και με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα συστήματα αντίστοιχα που ισχύουν σε άλλες χώρες όπως το Έστας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και έγινε και ακρόαση, ήρθαν συμπειρογνώμονες οι οποίοι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους μέχρι τώρα και είδαμε και σε ποιο βαθμό είναι συμβατά αυτά όλα που προτείνουμε σε τεχνικό επίπεδο με το EU LISA. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές τοπολογίες. Καταρχάς, προβλήματα εφαρμογής. Προσπαθούμε να αποφύγουμε, ακούγεται λίγο τεχνικό, αλλά είναι πολύ σοβαρό θέμα αν δεν αλλάξουν κάποια σημεία της πρότασης, προτείνεται πιο λεπτομερείς κανόνες για να καθοριστεί η χώρα η υπεύθυνη για την αξιολόγηση αιτιάς και την δυνατότητα να εφεσιβάλει ο ενδιαφερόμενος στην συγκεκριμένη διοικητική απόφαση, κάτι το οποίο θα καθορίζει επίσης και τις ευθύνες των κρατών για την σύνταξη αν θέλετε και τη συμμετοχή στο σύστημα προειδοποίησης για να μην δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα στις ομαδικές μετακινήσεις. Το σύστημα αυτό σε μια πρώτη φάση δεν θα ισχύει αυτού του είδους. Η σύνδεση με το αίτιας θα πρέπει να γίνεται μέσω μίας ηλεκτρονικής θηρίδας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωση και έβρεση πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αίτιας. Θα πρέπει οι υποψήφοι να ενημερώνονται για τη χρονική διάρκεια της άδειας και θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου συστήματος με δίκαιο τρόπο πρόταση προσπαθεί λοιπόν, οι προτάσεις που κάνουμε εμείς, να υπάρξουν περισσότερες ρήτρες εγγύησης για τους ταξιδιώτες και μεγαλύτερη ευκολία στην λειτουργία του συστήματος, να απαιτούνται έλεγχοι, να μην λειτουργεί με αυτοματισμούς ανεξέλεγκτους το σύστημα όταν οδηγεί σε αρνήσεις χορήγησης ε, θεώρησης θα πρέπει να ελέγχονται ανεξαρτήτως ε, του, της χώρας που γίνεται ο έλεγχος, οι τρόποι με τους οποίους ε, λειτουργεί η αστυνομική η συνοριακή αρχή και εφαρμόζει το σύστημα Θα πρέπει επίσης οι συνοριοφύλακες να έχουν την δυνατότητα πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα αιτιάς έτσι ώστε να κάνουν ένα έλεγχο δευτέρου επίπεδου αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο συνολικότερο. Είναι απαραίτητη η πρόσβαση αυτή έτσι ώστε η απόφαση την οποία θα λάβουν να είναι μια σωστά τεκμηριωμένη απόφαση. Υπάρχουν επίσης τροπολογίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να αποφεύγονται επικαλύψεις με άλλα συστήματα συλλογής πληροφοριών, να προστατεύονται επίσης μέσω του σωστού σχεδιασμού τους τα συστήματα αυτά από εξωτερικές προσβάσεις ή παραβιάσεις, να υπάρχει ανάληψη ευθύνης ελέγχου για την χρήση των στοιχείων αυτών, Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Είμαι βέβαιη ότι οι τροπολογίες σας έχουν σαν στόχο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία γύρω από ένα κείμενο το οποίο δεν είναι μόνο σωστού σκοπού αλλά και ένα κείμενο λειτουργικά θα έλεγα αποτελεσματικό. Αυτός είναι ο βασικός στόχος τον οποίο έχουμε και γι' αυτό προχωρούμε στην τροπολόγησή του και εύχομαι να συνεχίσω και ευχαριστώ και με, για τη μέχρι τώρα συνεργασία του συντονιστές. Κύριο Σίμονς τώρα έχει το λόγο από την, από την Κοινωνική Επιτροπή, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και θα ακούσουμε με ενδιαφέρον αυτά που θα μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κυρία Εισηγήτρια. Χαίρομαι που καταφέραμε αυτή τη φορά να συμπεριληφθεί ε, και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Εργασίας σας, που είναι ένα όργανο ε, που γνωμοδοτεί επίσημα και είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Και εγκαίρως ε, καταφέραμε να σας διαβιβάσουμε μια γνωμοδότηση που ψηφίστηκε ομόφωνα. Και μάλιστα ήρθε εγκαίρως και η μορφή. Φαίνεται ότι είναι αγαστή αυτή η συνεργασία μας. Και έχετε συμπεριλάβει και πολλά σημεία από τα όσα σας προτείναμε. Πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτή καθ' αυτή τη γνωμοδότηση και μετά μερικά σημεία που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί και να εστιάσουμε περισσότερο για να μην ε, ε, χαθούν από το σχέδιο έκθεσης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υπήρξε προβληματισμός για το αν υπάρχει καν ανάγκη για ένα σύστημα αίτιας. Ως εισηγητής κατέληξα σε μία διατύπωση που λέει το εξής. Το σύστημα αίτιας αυτή τη στιγμή είναι εκ των όν ουκάνευ, όχι απλώς αναγκαίο. Και κατά κατάφερα να πείσω τους συναδέλφους που ψήφισαν ομόφωνα την γνωμοδότηση εξηγώντας ότι όποιος αντιτίθεται σε ένα τέτοιο σύστημα αυτή τη στιγμή και καταψηφίζει θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του εάν έχουμε προβλήματα όταν έρχεται κάποιος από τρίτη χώρα. Αυτός είναι ένας από τους τρεις στόχους της γνωμοδότησής μας. Δεν το συνδέσαμε με προϋποθέσεις να συμπεριφθεί αυτό στο κείμενο της νομοθεσίας, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης, μιλούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, καμία διάκριση για την πρόσβαση στην εργασία και τα ε, λοιπά, όπως λέγεται και στην έκθεση του επόπτη για την προστασία των δεδομένων. Ε, μιλήσαμε και εμείς για τη διαλειτουργικότητα και τη διασυνδεσιμότητα για να μην υπάρχουν ε, διοικητικά εμπόδια. Και εσείς, όπως και εμείς, φροντίσατε πολύ περισσότερο από ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχετε και κάποια μέρημνα για τους πολίτες που δεν μπορούν να ζητήσουν ε, τη διαδικασία αυτή online επιγραμμικά. Ε, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και απαλλαγές, αλλά όλα αυτά μας βρίσκουν σύμφωνους και μας. Αλλά ένα τελευταίο που θέλουμε να πούμε και χρειάζεται προσοχή είναι η τελευταία παράγραφος, ε, η τελευταία πρόταση στην παράγραφο 3-4 όπου μιλούμε για αμοιβαιότητα ε, από τρίτες χώρες. Δηλαδή, σε περίπτωση που προβούν σε αντίπεινα κάποιες τρίτες χώρες, θα πέσουμε θύματα ε, κάποιων καταστάσεων και δεν θα μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί ελεύθερο στο Σέγγεν. Ε, κάποιοι άνθρωποι που θέλουμε να κυκλοφορούν. Τι γίνεται με το κόστος των ενδιαμέσων σε τρίτες χώρες. Ποιος θα το ελέγχει αυτό. Στην παραγραφο 4.3 στο τέλος το λέμε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα από τις αντιπροσωπείες, τις αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τρίτες χώρες λέτε. Αλλά στην πράξη δεν πηγαίνουν πάντα καλά τα πράγματα και ξεφεύγει το κόστος. Και τελικά μπορεί κανείς να θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει πρόθεση να ακριβίνει το κόστος για εκείνους που θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ορισμός των κριτηρίων για ε, κατηγορίες που εξαιρούνται. Παράδειγμα, το διπλωματικό προσωπικό Θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο περισσότερο. Προηγουμένως συζητήσαμε, Πρόεδρε, για ε, ποιοι είναι αυτοί που εκτελούν ε, αυτές τις πολιτικές. Εγώ συχνά έρχομαι στην Επιτροπή Μεταφορών Ε, υπάρχουν κάποιες μεταφορικές εταιρείες ε, που στην Επιτροπή Μεταφορών είναι σαφής ε, ο ορισμός αν πρόκειται για ξηρά θάλασσα ή αέρα. Αν θέλετε να το περιορίσετε στη θάλασσα και στον αέρα, τι γίνεται με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Την έχετε ξεχάσει στην πρόταση και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό μας απασχόλησε μας και ξέρω εκ πείρας ότι στο Δούναβι υπάρχει μεγάλη κίνηση κρουαζιέρας, κυρίως Αμερικανών. Ας πούμε που πάνε στη Σερβία και κάνουν κρουαζιέρα στο Δούναβι και κάποια στιγμή μπαίνουν και στη ζώνη Σέγγεν. Και υπάρχει μια εξαίρεση να μην φέρει την ευθύνη η εταιρεία ε, μεταφοράς. Ε, αλλά αυτό θα πρέπει να έχουμε ίδια κριτήρια για όλους και για τις χερσαίες μεταφορές και για τα αυτοκίνητα, για τα λεωφορεία και για το σιδηρόδρομο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πριν ε, δώσω το λόγο στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε πρώτα το λόγο στους και ηγητές ε, και τους συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν, διότι μπορεί να έχουν κάποιες ε, προτάσεις και ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Πρώτα λοιπόν οι σκιώδεις συγητές, η κυρία Ζίπελ θα μιλήσει εξ ονόματος της κυρίας Γκυγιόμ. Να σας δώσει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς η Σιλβίκη Γιόμ δεν μπορεί να παρευρεθεί λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων, αλλά μου έδωσε τις σημειώσεις της, τις οποίες και θα σας διαβάσω. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω τα θετικά της έκθεσης κυρίας Γκάλ. Ως εισηγήτρια, η κυρία Γκάλ διοργάνωσε Αρκετέ τεχνικέ συνεδριάσει με του και ηγητές στην Επιτροπή και άλλου ενδιαφερομένους για το σύστημα αιτία. Αυτό μα επέτρεψε να κατανοήσουμε καλύτερα την πρόταση και επομένω θα ήθελα να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Όσον αφορά την έκθεση, υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ενισχύει τι πληροφορίε που θα πρέπει να λαμβάνουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών ε, για την αίτηση και την έγκριση για τη διαδικασία ε, αιτίας. Ε, θέλει να εξασφαλίσει ότι ε, ένα θετικό ε, στοιχείο στην βάση δεδομένων της Interpol δεν σημαίνει απαραίτητα άρνηση εισόδου. Επίσης, ε, θέλει να υπάρχει εξασφάλιση και για τους ενδιαφερομένους. Προτείνει και ένα νέο σύστημα το οποίο θα καθορίζει ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση. Αυτό ε, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα τα διάφορα καθήκοντα που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη και να είναι και βέβαια τα κράτη-μέλη όταν ε, δημιουργούν σήμα ε, για κάποιον υπήκο της χώρας. Θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με κάποιον όταν υποβάλλει αίτηση για έγκριση στο σύστημα αίτιας. Κατά την άποψή μου όμως δεν αρκούν αυτά, πρέπει να γίνουν και άλλες τροποποίησεις του συστήματος, γι' αυτό και θα υποβάλω τροπολογίες κυρίως όσον αφορά την ε, ε, αρχή της μη διάκρισης και το profiling. Η γνωμοδότηση στη μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, λέει ότι μπορεί να υπάρξει de facto διάκριση και profiling μέσω της πρότασης αιτίας και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη η διαγραφή κάποιων στοιχείων που ζητούνται από τους υπηκόους ε, τρίτων χωρών, γιατί δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αν ζητήσουμε αυτά τα στοιχεία ε, είναι απαραίτητα ή αναλογικό. Επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι αρκετά θολά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως τα βασικά στοιχεία του συστήματος αιτιάς, ε, τους κανόνες ελέγχου και το σύστημα παρακολούθησης, τον κατάλογο μάλλον παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ρύθμιση ε, και τελευταίον, για να λειτουργεί ομαλά το σύστημα, ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν και πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποτίθεται ότι θα πρέπει να εξαιρούνται από τη θεώρηση διαβατηρίου. Αυτά είναι τα σχόλια από την Σιλβίκη Γιώμα. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια που αφορούν α, ε, όσα ακούσαμε μόλις από τον κύριο Σίμονς ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιον ο οποίος ε, ε, διασχίζει τα σύνορα και μετά έχουμε μια επίθεση. Συγγνώμη, αλλά με εκνευρίζει μια τέτοια δήλωση. Διότι οι επιθέσεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαπράχθησαν από άτομα τα οποία απλώς πέρασαν τα σύνορα και την επόμενη ή τη μεθεπόμενη διέπραξαν μια επίθεση. Οι επιθέσει έγιναν από ευρωπαίου πολίτε. Επομένω, ε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι έρχεται να προσθέσει όλο αυτό. Και όταν αναφέρεστε σε τρομοκράτε ε, και εγκληματίε, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί στι αρχέ, για αυτού ούτω ή άλλω υπάρχουν βάσει δεδομένων και δεν χρειάζεται το νέο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ζήπελ. Και ευχαριστώ και για τα σχόλια της κυρίας Κιγιόμ. Η κυρία Στίβενς τώρα, παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς φυσικά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και χαίρομαι που διαβάζω ότι γενικά υποστηρίζει την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης προτείνει να έχουν άμεση πρόσβαση και οι συνοριοφύλακες στο ΕΤΙΑΣ κατά τη διάρκεια του δευτέρου ελέγχου. Ενδιαφέρουσα γνώμη αυτή και η εναλλακτική λύση, εάν οι συνοριοφύλακες βλέπουν ως απόφαση μόνο ναι ή όχι από το σύστημα και δεν δεσμεύονται καθόλου από το σύστημα αυτό, ε, προφανώς μπορεί να χρειάζεται επιπλέον πληροφόρηση. Σε ό,τι αφορά δύο από τις τροπολογίες έχω κάποιες επιφυλάξεις η αρχική πρόταση με κάπως νεφελώδες και φέρει ότι ο δικαστής είναι εκείνο που αποφασίζει κατά πόσες αστυνομικέ αστυνομικές θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα και η συγγήτρια θέλει να αντικαταστήσει το δικαστή από κάποια κεντρική αρχή εντός εισαγωγικών. Αυτό μήπως στρέφεται κατά της αυτονομίας των κρατών μελών ε, για το πώς ε, ορίζουν και κανονίζουν την οικονομία τους. Και υπάρχουν και κάποιες εταιρείες ε, ταξιδιωτικά γραφεία που διοργανώνουν ταξίδια με λεωφορεία ή με το σιδηρόδρομο και ξερούνται από τη ρύθμιση αυτή. Νομίζω είναι υπερβολικό να ζητούμε να υπάρχει αυτή η έγκριση όταν κάποιος κυκλοφορεί με λεωφορείο ή με σιδηρόδρομο. Υπάρχει μια πρόταση που προτιμώ που είναι για το PNR το ευρωπαϊκό και το οποίο καλύπτει και τα λεωφορεία και το σιδηρόδρομο. Δηλαδή, να ζητούν απλούστατα από τον κόσμο να δείχνει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τις ταυτότητες αστυνομικές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και οι προλαλήσατες, θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την ποιότητα του προπαρασκευαστικού σας έργου που μας επέτρεψε να ε, παρουσιάσουμε ιδιαίτερα διαφορετικές απόψεις ε, για τα στοιχεία που λάγαμε, ε, για το περιεχόμενο και τους κινδύνους που ενέχει η πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ποιότητα όλης αυτής της προπαρασκευαστικής δουλειάς. Να σας πω ε, καταρχάς ότι η ομάδα μου υποστηρίζει την πρόταση, η οποία στόχο έχει να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και έγκρισης για τα ταξίδια. Βεβαίως, όπως και σε όλα τα μεγάλες κλίμακα συστήματα πληροφοριών, μία από τις πρώτες απαιτήσει είναι να υπάρχει μία αυστηρή ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων ασφαλείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και από αυτήν την άποψη υπάρχουν δύο λεπτά θέματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να καθορίσουμε σωστά τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουμε τους παράγοντες κινδύνους βάσει των οποίων θα συγκρίνονται τα στοιχεία του ετούντος. Ε, αυτά τα στοιχεία και οι δείκτες κινδύνου όσον αφορά την νόμιμη μετανάσταση και τη δημόσια υγεία θα πρέπει να διευκρινιστούν, λέει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κατάλληλα στοχευμένα και αναλογικά και αυτό φυσικά είναι και βασικό στοιχείο της δικής μας της ε, ευθύνης. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε επί του θέματος αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αιτιά που θα περιλαμβάνει κάποια ε, στοιχεία σας τα παραθέτω ουσιαστικά λέξη προς λέξη, ε, άτομα τα οποία είναι ύποπτα για διάπραξη σοβαρών ε, αδικημάτων και που θα μπορούσαν να διαπράξουν κάποιο άλλο έγκλημα ή αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε αυτός ο κατάλογος ε, παρακολούθησης να, είναι, ε, να χρησιμοποιείται καταλήλως από τα κράτη-μέλη και να εξασφαλίζουμε ότι όντως θα πρόκειται για άτομα τα οποία αποτελούν ε, υπαρκτό κίνδυνο σε θέματα ασφαλείας ή σε θέματα παράνομης μετανάστευσης. Κατά την άποψή μας λοιπόν θα πρέπει να ενισχύσουμε τις διάφορες εγγυήσεις και θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται και τακτική αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο ε, αξιολογούνται όλα αυτά τα κριτήρια κινδύνου. Και επίσης, ε, κάτι το οποίο θα πω και στη συνέχεια, δεν θα πρέπει ε, ο εκ των προτέρων έλεγχων, ε, έλεγχος των ατόμων που απαλλάσσονται από τη θεώρηση διαβατηρίων να είναι αυστηρότερος από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να παίρνουν θεώρηση διαβατηρίων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει περιορισμένη εδαφική έγκριση για το σύστημα αιτιάς. Ε, κατά την άποψή μας, οι 15 ημές και ο περιορισμός μόνο σε ένα κράτος μέλος ε, δεν είναι σωστός. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κατά πόσον μπορούμε να επιβάλλουμε τέτοιους περιορισμούς. Θα πρέπει επίσης, και θα επιμείνουμε από αυτού, ότι ο ετών θα πρέπει να γνωρίζει τους λόγους άρνησης και θα πρέπει να έχει και δικαίωμα άσκησης έφεσης σε περίπτωση που τους αρνηθεί ή ε, άδεια εισόδου ή αποσυρθεί η άδεια, ανακληθεί η αποσυρθει η ανακληθει εισόδου. Ε, όσον αφορά τη διάρκεια αυτής της έγκρισης, θεωρούμε ότι πέντε χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως θα πρέπει να περιοριστεί, θα μπορούσε να είναι δύο, τρία χρόνια είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν μέσα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα και επομένω ε, ε, μας απασχολεί αυτή η μεγάλη διάρκεια. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή από 5 σε 10 ευρώ. 5 ε, είναι φθηνότερο από ό,τι εφαρμόζουν όλες οι υπόλοιπε χώρες που έχουν ένα αντίστοιχο ε, σύστημα και ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Ξέρω ότι ε, ε, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πλούσιες και δεν θα έχουν τέτοιο πρόβλημα, αλλά ε, δεν μπορούμε να έχουμε τόσο χαμηλή τιμή. Θα μπορούσαμε να έχουμε υψηλότερη τιμή, να είμαστε στα 10 ευρώ, αλλά να αυξηθεί ο αριθμός των κατηγοριών που ε, δικαιούνται ε, δωρεάν τέτοια Παιδιά, ε, καλλιτέχνε ή άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν ω εκπρόσωποι μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπω για παράδειγμα γίνεται και με την πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίων. Θεωρούμε επίσης, όπως είπατε και εσείς ε, κυρία Πρόεδρε και κυρία συγήτρια ότι οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση, είτε πρόκειται για το δεύτερο έγγραφο, στις ε, έλεγχο συγγνώμη, στις πληροφορίες ε, που περιλαμβάνονται στο ΕΤΙΑΣ. Ε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε δυο φορές την ίδια δουλειά όταν υπάρχει ένα σύστημα μέσω του οποίου θα αρκεί μία καταγραφή και από εκεί και πέρα θα μπορεί κάποιος βάσει των στοιχείων αυτών να λάβει τη σωστή απόφαση. Υπάρχουν αρκετά βέβαια τεχνικά θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Τα αναφέρατε εσεί, δεν θα σταθώ εγώ στι λεπτομέρειε. Αλλά επιμένουμε ότι υπάρχει θέμα διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με άλλε βάσει δεδομένων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε και τι ε, θα μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι από ό,τι φαίνεται προσεχώς θα μας κάνει μια πρόταση. Στο έγγραφο δεν το είδα, ε, μπορεί και να το παράβλεψα εγώ, ε, δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για κάποια κράτη-μέλη που ακόμα δεν έχουν εφαρμόσει το κεκτημένο Σέγγερ πλήρω, ε, Βουλγαρία, ε, Ρουμανία, Κροατία και, ε, Κύπρος. Ε, αυτά λοιπόν κυρία Πρόεδρε από πλευράς μου. Well, uh, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις που πήραν μέρος στην συζήτηση που γίνεται σε αυτή τη φάση να σχολιάσω αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο εντελώς εκτός θέματος το να πει κανείς ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα προέρχονται από το εξωτερικό και διαπράχθησαν από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ξαναπατήσει το πόδι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι βέβαια σωστό και δεν είναι επίσης σωστό ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ήρθαν προήλθαν μερικές φορές από χώρες με εξαίρεση υποχρέωσης χορήγησης θεώρησης. Και ακόμα παραπάνω είπατε ότι όποιος είναι κατά του συστήματος αιτιάς θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τις μελλοντικέ επιθέσεις. Αυτή είναι μια σοβαρή ύβρις και μειώνει την αξιοπιστία του Ιδρύματός σας, του οργάνου σας. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση αυτή για το σύστημα αιτιάς την κάνουμε μακράν των δεδομένων και των γεγονότων. Είχαμε μία μελέτη των υπηρεσιών μας εδώ στο Κοινοβούλιο, η οποία στα ευρήματά της λέγει ότι συνολικά η αναγκαιότητα του αιτιάς δεν έχει τεκμηριωθεί. Λέγει η μελέτη των εμπειρογνωμόνων λέει ότι η ανάγκη που υπάρχει για τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και για τις στοχευμένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση ε, χορήγησης θεωρήσεων δεν έχει τεκμηριωθεί. Η αναγκαιότητα λοιπόν για ένα σύστημα το οποίο στοχεύει σε ταξιδιώτες από, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες με απαλλαγή είναι κάτι το οποίο δεν είναι και αυτό τεκμηριωμένο. Συνεπώς λοιπόν είναι λάθος να αναζητούμε αυτούς τους ανθρώπους. Όσοι προέρχονται από χώρες οι οποίοι έχουν εξαίρεση στον τομέα των θεωρήσεων, διαρωτάται κανείς ποιος είναι ο στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας. Όταν κάποιος θέλει να ζητήσει απαλλαγή από την χορήγηση θεώρησης στην Ένωση και το ψηφίσαμε εμείς αυτό, είναι απαραίτητο οι αστυνομικές αρχές της συγκεκριμένης χώρας να συνεργάζονται να ανταλλάσσουν σαν παράδειγμα πληροφορίες για γνωστούς ποινικού και ε, άλλους και άλλες κατηγορίες. Έχουμε το σύστημα Schengen και οι πληροφορίες αυτές τροφοδοτούν το σύστημα Schengen εφόσον οι διάφορες χώρες μέλη και οι χώρες που συνεργάζονται κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Οπότε αν κάποιος είναι εκτός του συστήματος οφείλουμε να το ελέγξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται εδώ να πούμε κάτι παραπάνω. Το σύστημα που προτείνεται είναι έτσι και αλλιώ πάρα πολύ ακριβό. Μισό δις υπολογίζεται το κόστος και είναι κάτι το οποίο παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα των ε, ε, ταξιδιωτών από τις χώρες αυτές. Η δημιουργία αυτής της τράπεζας δεδομένων μέσω της χονδρικής συλλογής προσωπικών χαρακτηριστικών είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δημιουργεί ε, μια σωρία ε, προσωπικών δεδομένων τα οποία θα παρακρατούνται χωρίς ε, καμία εξήγηση και δικαιολογία. Η συζήτηση για τα μέτρα αυτά μέχρι τώρα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Βασιστήκαμε σε φήμες ε, είπαμε ότι συλλέγοντας περισσότερα στοιχεία και παρεμποδίζοντας τον ερχομό ε, μιας κατηγορίας ανθρώπων θα πετύχουμε βήματα θετικά στον τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αυτό είναι λάθος. Ας πάρουμε μαθήματα από την ιστορία. Ε, καταρχάς να πούμε ότι η μετακίνηση ενός πολίτη είναι κάτι το αρχικά θετικό γιατί δίνει τη δυνατότητα από δημοκρατικές χώρες, ε, ε, σε πολίτες από δημοκρατικές χώρες να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να καταστήσουμε τη μετακίνηση αυτή ε, δύσκολη και ανέφικτη. Λυπάμαι αν το κάνουμε αυτό. Γιατί δυστυχώς εκεί φαίνεται να οδηγεί η συγκεκριμένη συζήτηση να οδηγεί δηλαδή σε ένα νομικό σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο αλλά αντιφάσκει θα έλεγα με την αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων που εφαρμόζεται και στους υποψήφιους ταξιδιώτες. Συνεπώς λοιπόν εγώ θα ήθελα να επανεξετάσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συζήτηση του συστήματος αυτού, του γιατί είναι απαραίτητο ένα τέτοιο σύστημα, αν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις πιο αποτελεσματικές και πιο στοχευμένες, τα χρήματα αυτά τα οποία θα πετάξουμε σε ένα τέτοιο σύστημα να τα επενδύαμε σαν παράδειγμα σε μέτρα καταστολήσει αστυνομικά μέτρα για τη συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές και από τις χώρες εξαιρέσεων υπό την καταδίγηση της Europol. Αυτά τα μέτρα θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά και στον τομέα της ασφάλειας και στον τομέα της καταπολέμησης των απειλών ε, εις βάρος της κοινωνίας μας και δεν χρειάζεται να συλλέγουμε άλλα προσωπικά στοιχεία όπως αυτά τα οποία προτείνει και γι' αυτό εξεπλάγει κύριε Ντεπρέ γιατί η πολιτική σας ομάδα όχι μόνο πολεμά υπέρ ενός τέτοιου συστήματος αλλά ζητά και τη διεύρυνση τη ε, της εμβέλειάς του. Ξέρω ότι είμαστε πλέον μια μειοψηφία γύρω από το θέμα αυτό αλλά δεν μπορούμε να μην συζητάμε τα πραγματικά τα γεγονότα και να αγνοούμε την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπρέ θέλει κάτι να σχολιάσει, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω μόνον ότι αν με είχε ακούσει προσεκτικά ο φίλος, εγώ αυτό το οποίο είπα στο πρώτο σημείο και σε αυτό που επέμεινα περισσότερο είναι ανάγκη ενίσχυσης των εγγυήσεων στους πολίτες και για τον καθορισμό του δίκτυ κινδύνου και για τον κατάλογο των ελεγχομένων και παρακολουθούμενων προσώπων. Εγώ είπα ότι υπάρχουν κίνδυνοι και πρέπει οι κίνδυνοι αυτοί να σταθμιστούν με σωστό τρόπο. Ε, δεύτερον, έρχομαι στην τελευταία σας πρόταση ότι δεν πρέπει να κάνουμε ένα ε, γενικό σύστημα, αλλά ένα επιμέρους σύστημα και να συνεργαστούμε με τις αστυνομικές αρχές ε, και τις συνοριοφύλακες των υπολείπων χωρών. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στον κύριο Ερντογάν. Αυτό θέλετε. Μην απαντήσετε τώρα, σας παρακαλώ. Έχουμε αρκετό χρόνο. Θέλουμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει. Μόνο την προσωπική ερώτηση. Αλλά θα, έχουν, ακολουθήσουν πολλές συνεδριάσεις σχεδόν, εδώ τον Ορίστε κύριε Άλμπραχτ. Σύντομος θα είμαι. Για το πρώτο σημείο μόνο. Δεν μπαίνω στο τελευταίο. Ε, σας ζητούν τα έγγραφα και τα στοιχεία όλων των ταξιδιωτών. Για εύλογους λόγους, αλλά στην αρχή ζητάτε όλα τα στοιχεία όλων των ταξιδιωτών και μετά γίνεται το φιλτράρισμα. Εγώ αυτό επικρίνω. Δεν είμαι βέβαιος ότι ανταποκρίνεται στα ζητή η απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει να έχει ειδοποιήσει πρώτα τον κίνδυνο και μετά να ζητά τα δεδομένα, όχι αδιακρίτως. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας και τη θετική σας στάση απέναντι στην εισηγήτρια. Βέβαια, παραμένουν πολλά ερωτηματικά. Να δώσω το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκρινίσει ορισμένα πράγματα και μετά στην Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε, καλησπέρα σα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Θέλουμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για τις προσπάθειες και την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ε, ως συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί ε, γενικώ. Καλωσορίζουμε την έκθεση. Το κείμενο παραμένει στο πνεύμα της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλαμε οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε κάποια σημεία που ίσως χρειάζεται συζήτηση. Το πρώτο ε, αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα αίτια των συνοροφυλάκων, λέει ο κύριος Θα πρέπει να μελετηθεί αυτό σοβαρά και ως προς την αναλογικότητα και ως προς τη σκοπιμότητα και να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο για εκείνους τα στοιχεία που χρειάζονται για να κάνουν τον έλεγχο στη δεύτερη φάση των ταξιδιωτών. Το δεύτερο αφορά τα ε, έσοδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ε, το τέλος που επιβάλλεται θα πρέπει να χαρακτηρίζεται εξωτερικό ε, εισόδημα ενώ το κείμενο της εισηγήτριας προτείνει ναι, ε, είναι εσωτερικευμένο αυτό το εισόδημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι ήταν, θα ήταν σκόπιμη μια τέτοια αλλαγή, διότι σε περίπτωση που έχουμε πλεόνασμα θα μπορούσαμε, αν είναι εξωτερικό το έσοδο, να παραμένει ε, το Ταμείο εσωτερική ασφάλεια και να χρησιμοποιηθεί τα επόμενα χρόνια, να μεταφέρεται από έτο σε για να ενισχυθεί ενδεχομένως ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων. Ε, πάση περιπτώσει, είτε είναι εσωτερικό είτε εξωτερικό το έσοδο αυτό. Στην προγραμματική περίοδο που βλέπει το εκάστοτε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αυτό το ποσό θα επιστρέψει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και άρα θα μειώνεται η εθνική συνεισφορά. Για τη Europol υπάρχουν κάποιες τροπολογίες της εισηγήτριας. Θα θέλαμε να τονίσουμε μόνο ότι η Europol δεν έχει άμεση πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών αιτίας και στα δεδομένα. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια. Η Europol δεν πρόκειται να έχει πρόσβαση σε καμία φάση της διαδικασίας. Προφανώς παραμένουμε στη διάθεσή σας για να υποστηρίξουμε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο και να σας βοηθήσουμε αν χρειάζεται να εξηγήσουμε διάφορα τεχνικά στοιχεία της πρότασης. Αν το θεωρείτε σκόπιμο. Η Επιτροπή ε, Πολιτικών Ευθύνων. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σουλών. Και τώρα για την Προεδρία του Συμβουλίου, η κυρία Άλισον Γκάτ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, η πρόταση αιτιάς ε, είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν το Συμβούλιο. Όπως είπατε και εσείς, ε, είναι σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πιο έξυπνο και πιο ισχυρό σύστημα πληροφοριών για την ασφάλεια συνόρων, τα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν ε, ένα τέτοιο σύστημα στον χάρτη πορεία τη Πρατισλάβα και ξανά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2016. Έκτοτε παρουσιάστηκε πρόταση τον Νοέμβριο, ξεκίνησαν οι εργασίες σε τεχνικό επίπεδο και μάλιστα αρκετά εντατικά και με τη συνεργασία όλων και την επικοδομητική προσέγγιση των κρατών μελών έχουμε πλέον τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων στις 9 Ιουνίου. Καλωσορίζω το σχέδιο εκθεσής σας κυρία Συγγήτρια και τα σχόλια που ακούστηκαν εδώ. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ε, έχετε κι εσείς μια γενική προσέγγιση, την οποία θα πρέπει ε, να τη συζητήσουμε και εντός του Συμβουλίου. Αλλά ε, πολλά από τα σημεία που έχετε επισημάνει κι εσείς είναι θέματα τα οποία και εμείς ε, συζητήσαμε και μάλιστα αρκετά εκτενώς και αντανακλώνται και στο κείμενό μας. Το αυτό ισχύει και για κάποια από τα σχόλια που ακούσαμε εδώ σήμερα από κάποιους βουλευτές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το μόνο που θα πω είναι ότι χαίρομαι και πάλι για το σχέδιο εκθεσή σας. Ε, περιμένουμε και να λάβετε τη διαπραγματευτική σας εντολή ώστε να ξεκινήσουν ε, οι διοργανικές διαπραγματεύσεις και εμείς από πλευράς μας, ε, δεδομένου ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο αυτό και τα όσα αναφέρονται και στην κοινή μας δήλωση. Προσβλέπουμε λοιπόν στις περαιτέρω συζητήσεις ε, και φαντάζομαι ότι αυτό θα κάνει και η μελλοντική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Γκάτ. Και για να κλείσουμε λοιπόν τη συζήτηση ως εισηγήτρια θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις, για τις ενθαρρυντικές τους προτάσεις. Γνωρίζω ότι υπάρχει διάσταση απόψεων. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια κοινή θέση στο τέλος, ε, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι εύκολο. Όπως σας είπα και στην αρχή στην παρουσίασή μου, γνωρίζω ότι αυτή η έκθεση και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφήνει μεγάλο περιθώριο για βελτιώσεις, ε, διευκρινήσεις ε, και αυτή είναι και η δουλειά μας. Ε, πρέπει να βελτιώσουμε το κείμενο και να προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι το οποίο θα είναι και πιο εύκολο στην εφαρμογή του. Συμφωνώ πολύ με τον κύριο Ντεπρέ. Γι' αυτό άλλωστε το είπα και εγώ και έχω συμπεριλάβει και σχετική τροπολογία αυτοί οι οποίοι εξαιρούνται τη απαλλαγή θεώρηση διαβατηρίου δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε δυνότερη θέση και να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες ε, ε, για να ε, μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτούς που έχουν θεώρηση διαβατηρίου. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί και το κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρθηκαν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Είμαι βέβαιη ότι θα βρούμε απαντήσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω και συγκεκριμένες προτάσεις να σας κάνω και αντιλαμβάνομαι και πλήρως γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα και γιατί κάποια άλλα απουσιάζουν, αλλά ελπίζω ότι στη συνεδριάση των σκιωδών εισηγητών θα μπορέσουμε να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι με το σύστημα εισόδου-εξόδου ε, που έχουμε τώρα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σίγουρα θα επηρεάσουν και το θέμα αυτό. Επομένως, θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε και τι συμβαίνει με το σύστημα εισόδου-εξόδου για να μην βρεθούμε να έχουμε ε, διπλές ε, εργασίες στη συνέχεια. Όταν εγκρίνεται κάτι εδώ θα πρέπει να εξετάζουμε και τι γίνεται στο σύστημα εισόδου-εξόδου για να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τα ευθυγραμμίσουμε όλα αυτά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο σύστημα εισόδου-εξόδου. Η αρχική προθεσμία για τροπολογίες ήταν 11 Ιουλίου, αλλά η κυρία Βερζιά, η κυρία Γκυγιόμ και ο κύριος Άλπρεχτ μου ζήτησαν να παραταθεί η προθεσμία μέχρι τις 18 Ιουλίου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τροπολογίες και τη δέχομαι λοιπόν την πρόταση. Προθεσμία λοιπόν κατάθεση τροπολογιών 18 Ιουλίου, 4 Ιουλίου το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συνεργασία, περιμένω τις προτάσεις τροπολογιών σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς και θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα καλό κείμενο το οποίο θα είναι και βιώσιμο όταν θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην πράξη και να μην μείνουμε μόνο στα θεωρητικά. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Και τώρα. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης. Θα πρέπει να συζητήσουμε από κοινού τα επόμενα τρία σημεία. Την αποστολή της Επιτροπής Λιμπεστή Hot Spot στην Ελλάδα και στην Αθήνα 22 με 25 Μαΐου του 2017 την έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή της ε, δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, έκτη αναθεώρηση. Πρόκειται για κοινή συζήτηση λοιπόν για την κατάσταση στην Ελλάδα. Μια αντιπροσωπεία της ΛΥΜΠΕ επισκέφθηκε την Ελλάδα όπως σας είπα. Ο συνάδελφο Πίτερ Νίντορ Μίλλερ ήταν επικεφαλή αντιπροσωπείας και συμμετείχε και η κυρία Ελένη Θεοχάρου. Ο στόχο ήταν να δούμε το σύστημα υποδοχής στην Ελλάδα, καθώς επίσης και γενικότερα τη διαχείριση της μετανάστευση ε, βάσει και τη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και των hot Οι συνάδελφοι επισκέφθηκαν δύο hot spot ε, στην Κο και στη Λέσβο, καθώς επίσης και διάφορες καταστάσεις υποδοχής. Συναντήθηκαν με εκπροσώπους των ελληνικών αρχών, ε, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευρωπαϊκές υπηρεσίες, την υπατιαρμοστία των ΟΕΕ για τους πρόσφυγες το σχέδιο έκθεσης θα το παρουσιάσει τώρα ο επικεφαλής αντιπροσωπεία και μετά από την παρουσίασή του θα περάσω στα επόμενα δύο σημεία της κοινή συζήτηση. Μετά λοιπόν θα ακούσουμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 13η έκθεση για την ε, επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση από τον κύριο Νίλσεν. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Και στη συνέχεια την παρουσία του κυρίου Βερβέη για την εφαρμογή της ε, ε, δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η αντιπροσωπεία κατά την επίσκεψη στην Ελλάδα είχε σκοπό να σας συναντήσει, αλλά επειδή υπήρξαν και κάποιοι χρονικοί περιορισμοί, δεν κατέστη δυνατό. Είστε λοιπόν εδώ σήμερα και θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Να δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Νίτερ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η αποστολή στην Ελλάδα έλαβε χώρα από τις 22 μέχρι τις 25 Μαΐου. Και όπως ήδη είπατε κυρία Πρόεδρε, είχαμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα αυτό το τρίμερο. Επισκεφτήκαμε διάφορες εγκαταστάσεις, hot spots, προαναχωρησιακά κέντρα, ε, ε, στέγες ε, ασυνόδευτων ανηλίκων και στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Είχαμε πολλές συνεδριάσεις με ΜΚΟ, με εκπροσώπους των ελληνικών αρχών και φυσικά συναντήσαμε και τον Υπουργό Μετανάστευσης βάσει ε, αυτής της επισκόπησης που ήταν και πλατιά ε, της κατάστασης στην Ελλάδα σημείωσε κυρίως η αντιπροσωπεία τα εξής. Οι ε, συνθήκες υποδοχής στα hotspot και στις εγκαταστάσεις που επισκεφθήκαμε βελτιώθηκαν τους τελευταίους μήνες, ωστόσο παραμένει η ανησυχία ως προς τις συνθήκες που επικρατούν σε κάποιους καταβλισμούς. Δεύτερον, κάνει προσπάθειες η ελληνική υπηρεσία ασύλου να ενισχυθεί το σύστημα. Οι ελληνικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες συμπεριλαμβανομένες και με τη βοήθεια της ΙΑΣΟ ε, του Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου για να τηρούνται οι προθεσμίες. Ε, ωστόσο ακόμα δεν ε, τηρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές. Μεγάλη ε, είναι η καθυστέρηση και πάρα πολλοί ετούντε περιμένουν να διεκπαιρεωθούν οι φακελοί του για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμα που προκαλεί προβλήματα στα νησιά. Επίση, εκείνοι που δεν είναι επιλέξιμοι για διεθνή προστασία πρέπει να επιστρέφουν. Το πρόβλημα έχει οξυνθεί γιατί άλλαξαν οι μεταναστευτικέ ροέ τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα την περασμένη χρονιά. Στη συνέχεια, ε, η αλλαγή ε, του νομικού και θεσμικού πλαισίου ε, δυσκόλεψε περισσότερο και τους φορείς αλλά και τους ετούντες άσυλο για να ενημερώνονται ε, με σωστό τρόπο και να έχουν και νομική ε, βοήθεια ή τουλάχιστον νομική βοήθεια είναι περιορισμένη. Πέμπτον, η διαδικασία ταυτοποίησης ευάλωτων ομάδων κατά τη διάρκεια της υποδοχής θα πρέπει να συστηματοποιηθεί περισσότερο. Επόμενο θέμα, η σημασία ε, συνεχούς και βιώσιμης χρηματοδότησης ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε παρά να το τονίσουμε αυτό, γιατί τώρα σταματάει η έκτακτη χρηματοδότηση ε, και αυτό έχει πολύ ανετικές συνέπειες επιτόπου, ιδιαίτερα στα νησιά. Και ένα τελευταίο σημείο στην υπηρετική Ελλάδα φοιτούν τα παιδιά στο σχολείο και αυτό το αναγνωρίζουμε, αλλά στα νησιά είναι μεγάλο το πρόβλημα γιατί περιμένουν μεγάλε περιόδου μαζί με του γονεί του, ε, πριν είναι, να είναι σε θέση να έχουν ένα ε, μέλλον, να μορφωθούν και μήκυο ε, έχουν κάποιε δράσει, αλλά αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κανονικό σχολείο. Ανταλλάξαμε απόψει με όλου και κάναμε τι εξή συστάσει. Και η κυρία Βίνμπεργκ είναι εδώ. Η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται περιορισμένα μόνο για εκείνους που επιλέγουν την εθελούσια επιστροφή. Θα πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά τον κίνδυνο εξαφάνισης ε, των υποψηφίων, αλλά αυτό θα πρέπει να το ελέγχουν ανεξάρτητοι παρατηρητές. Επίσης, η πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση θα πρέπει να ε, εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ένταξη έτσι ώστε οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να έχουν την ευκαιρία να εντάσσονται στην κοινωνία που τους υποδέχεται και να γίνονται αποδεκτοί από τον τοπικό πληθυσμό. Επόμενη σύσταση, τέταρτη ταυτοποίηση οικογενειακών δεσμών και οικογενική επανένωση υπό τις διαδικασίες του Δουβλίου θα πρέπει να επιταχυνθούν. Και όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να συνεργάζονται προς τον σκοπό αυτό. Και τελευταία σύσταση, η μετεγκατάσταση πρέπει να επιταχυνθεί. Θα πρέπει να ε, πιεστούν τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τις ε, υποχρεώσεις τους βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου στην Ελλάδα υπάρχουν 12.000 ε, σήμερα ε, προς ε, μετακατάσταση. Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της και οι άνθρωποι αυτοί αναμένουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέλει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για τη μετακατάσταση και μετά τις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πραγματικά την αίσθηση ότι οι ελληνικές αρχές και η ελληνική κυβέρνηση κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά είδαμε ότι παραμένουν τα προβλήματα και μάλιστα πολλά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νίτερ Μιουλέρ. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, θα ήθελα να το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Νίλσον, για να μας παρουσιάσει τη 13η έκθεση για την ε, μετακατάσταση και την επανεγκατάσταση. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, πού βρισκόμαστε. 15.000 από Ελλάδα, επανεγκατάσταση και 7.000 από Ιταλία. Θετική η τάση, σημαντικές βελτιώσεις ιδιαίτερα από Ιταλία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη για την Ιταλία θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες αναλήψεις υποχρεώσεων από κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχουμε λιγότερο αυστηρές ρυθμίσεις, γιατί λειτουργούν σαν εμπόδιο στη διαδικασία και ζητάμε από όλους τους εμπλεκομένους να συντονίζονται σωστά έτσι ώστε να αποφεύγονται ε, προβλήματα ε, ταυτόχρονης σύμπτωσης στις μετεγκαταστάσεις από Ελλάδα και Ιταλία. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης σωστή καταγραφή όλων αυτών που είναι υποψήφιοι για επανεγκατάσταση να απλοποιηθεί η διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια. Ας έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία πληροφόρηση στην Ιταλία για την καταγραφή. Έχουμε δώσει οικονομική στήριξη έτσι ώστε η διαδικασία να είναι καλύτερη και πιο συγκεντρωτική επηρεάζοντας θετικά την ταχύτητά της. Νομίζω ότι θα πρέπει με τις συμπληρωματικές προσπάθειες να πετύχουμε τον κοινό στόχο, να μετεγκαταστήσουμε δηλαδή όλους αυτούς που είναι καταγεγραμμένοι στην Ελλάδα και την Ιταλία πριν από το τέλος της διάρκειας που προβλέπεται. Αυτό θα πρέπει όμως να γίνει μετά από προσπάθειες των κρατών μελών με δίκαιο τρόπο και αναλογικό τρόπο Ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάσης βάρος Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας. Δεν έχουν αναλάβει υποχρεώσεις, δεν έχουν μετεγκαταστήσει κανέναν τον τελευταίο 12 χρόνο. Όπως είπαμε... 15,500 persons resettled under the July conclusions. That's overall a positive development. Uh, τους τελευταίους 12 μήνες, τον τελευταίο χρόνο λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια κάποια λύση στο πρόβλημα. Θα πρέπει να το κάνουν έστω και την τελευταία στιγμή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονικά. Από την Τουρκία έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή ενημέρωση για 6.200 άτομα τα οποία έχουν επιστρέψει. Είχα ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση για την έκθεση, αλλά ίσως θα ήταν πιο ενδιαφέρον να σχολιάσω την έκθεση της Επιτροπής και μετά στο ενδιάμεσα θα μπορούσα να σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία ε, προκύπτουν από τη δική μας την έκθεση. Θα ήθελα καταρχάς ε, να σας πω ότι σε γενικές γραμμές ε, θεωρώ ότι η έκθεση, όπως παρουσιάστηκε, είναι αρκετά ισορροπημένη και βέβαια σε μεγάλο βαθμό Τίχνουν τα ίδια επιτολέσματα, την ίδια εντύπωση που έχουμε αποκομίσει και εμείς. Οι συνθήκες υπεδοχής έχουν βελτιωθεί αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες. Νομίζω ότι αυτό συνοψίζει πολύ σωστά την κατάσταση. Έχουν ε, υπάρξει σαφείς προσπάθειες ε, και από τις δύο πλευρές των συνόρων για βελτιώσεις. Ε, υπάρχουν βελτιώσεις, κυρίως σε σχέση με τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζαμε το χειμώνα. Βεβαίως εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωση και υπάρχουν και κάποιε ανησυχίε για συγκεκριμένα μέρη και θα ήθελα να σας πω μια συγκεκριμένη ανησυχία που εξακολουθώ να έχω και αφορά την κατάσταση στοιχείο, ιδίως στη στη Σούδα που δεν είναι επίσημος ο χώρος υποδοχής, ε, είναι κάτι το οποίο ε, είναι υπό την αρμοδιότητα του Δήμου, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων ε, και ήδη έχουμε προτείνει αρκετές άλλες λύσεις και χρηματοδότηση για άλλες λύσεις, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστούν οι κάτοικοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, και το θέμα έχει κολλήσει λοιπόν και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερως. Υπάρχουν και άλλες ανησυχίες, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ε, έχουμε διαπιστώσει βελτιώσεις. Αναφέρθηκε επίσης ότι... Ε, Υπάρχει θέμα με τις διαδικασίες. Ε, πρέπει να πω, για να διευκρινίσω την κατάσταση, ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδο σε επίπεδο υπηρεσιών ασύλου ε, και με την υποστήριξη της ΕΑΣΟ ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, διότι παρασχέθηκε υποστήριξη αλλά το πρόβλημα, και αναγνωρίζω και τη δική σας την απογοήτευση, έγκυται στο δεύτερο ε, στάδιο αποφάσεων, δηλαδή στη διαδικασία της έφεσης. Και προσφυγών. Και φυσικά ε, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε εμείς προσπάθεια. Ίσα ίσα διπλασιάστηκε ε, το προσωπικό για την ε, εξέταση των προσφυγών. Έχουμε και παροχή υπολογιστών, νομική συνδρομή. Έγιναν πάρα πολλά λοιπόν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά προς το παρόν δεν μεταφράζεται αυτό σε αύξηση του αριθμού υποθέσεων που διεκπεραιώνονται. Και μεγάλος αριθμός αυτών των υποθέσεων δεν είναι πρόσφυγες ε, αυτοί καθ' αυτή, αλλά είναι μάλλον άτομα που κατά πάσα πιθανότητα δεν δικαιούνται διεθνού η προστασία. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι δύσκολο να υπάρξει πρόοδος για την επιστροφή τους είναι ακριβώς ε, επειδή ε, δεν θεωρούνται πρόσφυγες. Και φυσικά αυτό παρακολουθεί το όλο σύστημα. Ε, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την αναγνώριση κάποιων αδυναμιών και ε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω όμως ότι μέχρι τώρα το σύστημα Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα εντάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων. Και φυσικά οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στη συνέχεια είναι ότι θεωρούνται ότι εμπίπτουν σε συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα και αυτό φαίνεται και στα στατιστικά στοιχεία. Μέχρι τώρα πάνω από 8.000 άτομα ε, παραπέμπονται στην τακτική διαδικασία ακριβώ λόγω του γεγονότο ότι εμπίπτουν σε ευάλωτε ομάδες και αυτό φυσικά έχει ε, σημασία για, συνολικ... για τους συνολικούς αριθμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί παρούσα και θα συνεχίσει να είναι παρούσα για χρηματοδότηση. Αλλά ε, προς το παρόν η χρηματοδότηση που έχει παρασχεθεί ε, είναι κυρίως για κατεπίγουσα βοήθεια και μέσω και του μέσου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ και πάλι δηλαδή μέσω για κατεπίγουσα βοήθεια. Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση και να αρχίσει να χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση ε, του Εθνικού Κονδυλίου της Ελλάδος. Εξακολουθεί να είναι ε, χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο γιατί απαιτούνται και συγκεκριμένε δυνατότητες και η αλήθεια είναι, και γι' αυτό ε, έχουμε και αυτές τις καταγγελίες και τις ανησυχίες, οι εταίροι προτιμούν να έχουν ως ε, οικονομικό συνομιλητή τους ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το ελληνικό κράτος. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ε, να βοηθήσουμε τη διαχειριστική αρχή να κάνει τη μετάβαση, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε στενά το θέμα, διότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν θα πρέπει ε, να ε, σημαίνει αυτό ότι δεν θα είναι στο ίδιο ύψος οι υπηρεσίες ούτε στα νησιά ούτε στην ενδοχώρα. Παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση στενά. Κράτηση. Ε, μόνο ε, κατά περίπτωση και ως ίστατη λύση και εδώ συμφωνώ ότι για διάφορους λόγους υπάρχει και η ανθρωπιστική πτυχή, αλλά υπάρχει και μια πολύ πρακτική πτυχή για τις δυνατότητες κράτησης. Είναι πολύ περιορισμένες αυτές, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό. Και για τους δύο αυτούς λόγους ε, συμβουλεύουμε τις ελληνικές αρχές να μην ε, ε, μεταφέρονται υποψήφοι για ε, εθελοντική επιστροφή σε χώρους κράτησης. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πει ότι θέλουν να επιστρέψουν, ε, κατά εμάς δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται σε κέντρα κράτησης. Και για να σας δώσω και την όλη εικόνα, υπάρχουν κάποιοι νομικοί περιορισμοί που οδηγούν τις ελληνικέ αρχές στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει και είμαστε σε συνεχή συνομιλία επ' αυτού και αν μου επιτρέπετε εγώ θα έκανα αυτό που προτείνεται για την επανένωση οικογενειών ε, ε, Νομίζω ότι θα έπρεπε να τη δώσω σε εσά την ερώτηση. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτές οι διαδικασίες ε, γίνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η διαδικασία της ε, μετεγκατάστασης έχει ε, ήδη αναφερθεί. Έχουμε πει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις επ' αυτού. Και τέλος, ε, υπήρξε κάποιο σχόλιο για ε, τα παιδιά στο σχολείο και τη σχολική τους εκπαίδευση και την όλη διαδικασία ένταξης και τα σχετικά κονδύλια. Ε, συμφωνώ απολύτως με μια μικρή διαφορά. Πρώτο μας μέλημα θα έπρεπε να είναι να είμαστε βέβαιοι ότι η παραμονή των ανθρώπων στα νησιά θα είναι στο δυνατόν πιο περιορισμένη σε βαθμό δηλαδή που έχουμε και παιδιά να μην πρέπει να μείνουν παραπάνω από το απολύτως απαραίτητο στα νησιά ώστε να μπορούν ε, να ε, συμμετέχουν στο σχολείο, να πηγαίνουν σχολείο ε, στην χώρα. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμελούμε και τα παιδιά που βρίσκονται στα νησιά και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να αρχίσουμε να εξετάζουμε και τι θα γίνει στη συνέχεια. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε κάποια άλλα μέρη ή σε κάποια άλλα κρατημέλη, πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα. Επομένως, ε, τίθεται θέμα ένταξή τους. Ε, αυτό έχει αναγνωριστεί και ε, θα έλεγα ότι αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι από αυτού και επομένως σας ευχαριστώ πολύ για τη σύσταση. Και νομίζω ότι με αυτά σας είπα και λίγα πράγματα για το πού βρισκόμαστε με την εφαρμογή της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Νομίζω ότι αν εξετάσουμε τους αυστηρούς στόχους της δήλωσης ε, μπορούμε να πούμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε αποτελέσματα ε, και να εκπληρώνονται οι στόχοι, ο αριθμός των αφήξεων εξακολουθεί να είναι χαμηλός, εξακολουθούμε να έχουμε πολύ λιγότερους θανάτους στο Αιγαίο από ό,τι είχαμε στο παρελθόν, αλλά στο πρώτο επίπεδο τα πράγματα σίγουρα έχουν βελτιωθεί, υπάρχουν όμως ε, και ε, ε, πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και νομίζω ότι πολύ σωστά τα είπατε και εσείς στην έκθεσή σας εδώ στην Επιτροπή. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βέβε. Οι συνάδελφοι που πήραν μέρος στην αντιπροσωπεία δεν ξέρω αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Και μετά η κυρία Γκόμες. Spinelli? Okay. So, uh, Mrs. Ernst. Λοιπόν, ε, κύριε Ernst, πρώτη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση τόσο κοντά χρονικά μετά την αποστολή, γιατί είναι και απαραίτητη. Και σε μερικά σημεία δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν. Σε ό,τι αφορά το ταξίδι στην Ελλάδα, βελτιώθηκαν οι συνθήκες υποδοχής, ισχύει αυτό και φιλοξενίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που κυρίως έχουν να κάνουν με τη συμφωνία με την Τουρκία, τη λεγόμενη δήλωση και απορρέουν και από τη συμφωνία αυτή. Θα ήθελα να αφαιρθώ στα εξή θέματα και παρακαλώ να απαντήσετε. Πρώτον, κράτηση. Είπατε ότι η κράτηση ε, είναι μια απόφαση της Ελλάδας γιατί θεωρεί ότι φροντίζει καλύτερα εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν ε, εθελουσίες σε αυτά τα λεγόμενα προαναχωρησιακά κέντρα. Ξέρουμε πως είναι τα επισκεφθήκαμε. Είναι κλειστά κέντρα. Μπορεί κάποιος να βγει για κάποιο διάστημα, αλλά γιατί και ποιος το σκέφτηκε και με ποιο τρόπο ότι είναι τρία είδη των ανθρώπων και ζητώ συγγνώμη που το αναφέρω έτσι που πρέπει να κρατούνται εκεί. Εκείνοι που είναι ε, προς απέλαση, ε, εκείνοι που εθελοντικά θέλουν να επιστρέψουν και η τρίτη είναι δεχόμενη, ε, λεγόμενη παραβατική, αυτή που μας τους ανέφεραν ως trouble Και επανειλημμένα ακούσαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη απόφαση μετά την προσφυγή. Πώς έχει διαδικασία. Παίρνεις την πρώτη απορριπτική απόφαση και μετά θα πρέπει να αποφασίσεις αν θα επιστρέψεις ε, εθελοντικά ή όχι. Αν θέλεις να κάνεις προσφυγή, τότε δεν έχεις πια τη δυνατότητα ή μόνο περιορισμένη να επιστρέψει κανείς εθελοντικά για να έχει την ε, οικονομική στήριξη. Αυτό ποιος το αποφάσισε, η Ελλάδα. Ποιος ε, έλαβε αυτή την απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στηρίζει, την επιθυμεί, μήπως την έχει ορίσει κιόλας. Το τρίτο, οικογενειακή επανένωση είναι πάρα πολύ αργή αυτή η διαδικασία και τραβάει σε μεγάλο μάκρος και θα σας παρακαλέσω να μας πείτε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ποιες είναι οι αιτίες, πώς αντιδρούν τα κρατη δεν είναι πρόθυμα να δεχτούν την οικογενική επανένωση και να την προωθήσουν με ταχύτερους ρυθμούς. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που επικρατούν το τρίτο για τη μετεγκατάσταση 12.000 ε, εκκρεμούσαν, τώρα είναι 8.000 άνθρωποι που έχουν κάνει τις βαλίτσες τους. Ουσιαστικά κάθονται πάνω και περιμένουν να μετακατασταθούν. Αλλά τα κράτη-μέλη λένε ότι ε, δεν ξέρω, δεν θέλουμε, δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χώρο, δεν μπορούμε να τους υποδεχθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει. Γιατί περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί να μετακατασταθούν και δεν τους υποδέχονται. Για τα χρήματα είπατε όταν φύγει η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ θα πρέπει αυτό να καλύπτεται από εθνικού πόρους. Και πώς γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Για ένα τελευταίο. Τι γίνεται με τις ευάλωτε ομάδες. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας νόμος στην Ελλάδα για να έχουν ειδική υποστήριξη, να μην στεγάζονται στα κέντρα φιλοξενίας και υποδοχής. Μάθαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί πιέσει να μην εφαρμοστεί ο λαγονόμος με τον τρόπο αυτό. Και αυτές οι ευάλωτες ομάδες ε, να μπορούν να επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Ε, για τα παιδιά στα σχολεία. Στη Μόρια υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν και 10 και 11 μήνες και δεν υπάρχει σχολείο για τα παιδιά. Υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ που τα απασχολούν με ε, κάποια προγράμματα ψυχαγωγίας κτλ. Γιατί δεν ε, μεταφέρονται οι άνθρωποι αυτοί στην επιρωτική Ελλάδα. Ευχαριστώ κυρία Γουίνμπεργκ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε πήρα και εγώ μέρος σε αυτή την μετάβαση στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους οργάνωσαν το είναι επίσκεψη αυτή, η οποία είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα. Ιδιαίτερα ειδωμένη από την πλευρά μιας Σουηδής. Εμείς φυσικά δεν στείλαμε μετανάστες στην Ελλάδα. Ε, υπήρξαν όμως μετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα από άλλες χώρες και κατέληξαν στην Σουηδία Μας είχαν πει στην Σουηδία ότι το σύστημα υποδοχής ήταν πάρα πολύ κακό, αλλά εγώ ε, θα έλεγα ότι εντυπωσιάστηκα θετικά από αυτά που είδα στην Ελλάδα. Ε, υπήρχαν χώροι πολιτισμένοι με κλιματισμό, με δορυφορικές κεραίες, υπήρχαν γιορτές με μπάρμπεκιου, ε, πραγματικά εγώ δούλευα σε ταξιδιωτικό γραφείο και πούλησα κάποιες εκδρομές για χρόνια σε μέρη λιγότερο θα έλεγα πολυτελή από αυτά. Οπότε τώρα κανονικά θα έπρεπε να πάω στη Σουηδία και να πω ότι μπορούμε να τους ξαναστέλνουμε στην Ελλάδα γιατί οι συνθήκες δεν είναι κακές. Οι υπεύθυνοι τώρα που συναντήσαμε στην Ελλάδα, υπουργό αρχές αστυνομικές κτλ. μας είπαν ότι άνω το 80% των προσφύγων στην Ελλάδα ή μάλλον αυτών που ήταν στην Ελλάδα ήσαν οικονομικοί μετανάστες. Δεν υπάρχουν πραγματικοί δηλαδή ετούντε άσυλο. Πρόκειται για ανθρώπους που προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές όπως και τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι κυρίως οι οικονομικοί μετανάστες. Αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα μακροχρόνιες. Μίλησα με αυτούς που ζουν σε αυτά τα κέντρα υποδοχής, μίλησα με αυτούς που ήξεραν ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν στην Τουρκία και ότι έπρεπε να περιμένουν πάρα πολύ καιρό πριν γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι χρονοβόρο σαν διαδικασία και δημιουργεί προβλήματα και αυτό με ανησυχεί. Ήμασταν σε ένα κέντρο υποδοχής στη Λέσβο συναντηθήκαμε αν δεν κάνω λάθος με οκτώ άνδρες από τη Βόρεια Αφρική οι οποίοι μας περιέγραψαν την κατάστασή τους. Μας είπαν ότι το Wi-Fi ήταν μαύρα χάλια. Η τροφή ήταν ε, κακή, ούτε για σκύλους. Και ταυτόχρονα άρχισαν να μου λένε ότι αν δεν έπαιρναν αμέσως άσυλο στην Ελλάδα, τότε σε αυτή την περίπτωση είτε θα έφευγαν κρυφά στην υπόλοιπη χώρα ή θα ξεσπούσαν σε πράξεις βίας. Και αυτό βέβαια μου έκανε τρομερή εντύπωση. Uh, Ευχαριστώ κυρία Βίνμπεργκ. κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας, αλλά διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση. Το Κοινοβούλιο πραγματικά πολύ καλά έκανε να πάει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση έχουν βελτιωθεί πολλά σε ό,τι αφορά την ποιότητα των κέντρων υποδοχής. Και αυτό πραγματικά αντιστοιχεί στη γενεοδορία και στην αλληλεγγύη που έχει δείξει ο ελληνικός λαός απέναντι στους πρόσφυγες. Στην έκθεση αυτή όμως διαπιστώνω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια κακό κείμενα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Τα παιδιά αυτά έχουν ε, πρόβλημα επιτροπίας. Δεν υπάρχει κάποιος που να ασχολείται ε, ουσιαστικά με αυτά τα παιδιά και η έκθεση λέει ότι 900 ανήλικοι έχουν εξαφανιστεί. Και έχουν εξαφανιστεί για λάθος λόγους, όχι επειδή βρήκαν την οικογένειά τους ή βρήκαν έναν τρόπο να ε, μεταβούν εκεί που ζει η οικογένειά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι τίθεται ένα ζήτημα ασφαλείας για όλους μας. Γιατί τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν πέσει θύματα δικτύων οργανωμένου εγκλήματος. Και επίση κάτι άλλο που με ανησυχεί είναι ε, τι γίνεται με την ε, δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας γιατί αυτό είναι τελείως ε, αμφιβόλου ποιότητας ως συμφωνία, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου και τη βοήθεια στους πρόσφυγες. Η έκθεση τα εξηγεί όλα αυτά πάρα πολύ παραστατικά. Πριν ε, κάνω την ερώτηση που έχω όμως θα ήθελα να πω ακόμα ότι χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους ανέλαβε δράση απέναντι στα κράτη-μέλη εκείνα που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την υποδοχή προσφύγων. Έχετε λοιπόν προβεί σε αυτή τη διαδικασία προσφύγηση παραβάση Ξέρω ότι είναι πολύ χρονοβέρες οι διαδικασίες. Δεν κατηγορώ την Ελλάδα. Ε, ξέρουμε ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες. Στην περίπτωση της μετεγκατάστασης υπήρξαν πολλές δευτερογενείς μετακινήσεις και γνωρίζω τι συμβαίνει ε, στην Πορτογαλία. Χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες που έχουν μετακατασταθεί από την Ελλάδα και την Ιταλία και περίπου 40%, 40 ε, ξαναφεύγουν και ε, πηγαίνουν στις χώρες που ήθελαν από την αρχή να καταλήξουν επειδή έχουν οικογένεια εκεί. Όσο ε, αφήνουμε τους ανθρώπους εγκαταλείπουμε στην Ελλάδα και στην Ιταλία για να περιμένουν μια λύση, τόσο πιο εύκολο είναι να πέσουν στα νύχια των δικτύων των διακινητών και να έχουμε δευτερογενείς μετακινήσεις προς άλλες χώρες. Είναι ένας φαύλος κύκλος και τελικά καταλήγουν στη χώρα που ήθελαν ε, να πάνε αρχικά, στη χώρα προορισμού, περνώντας από κάποιες άλλες χώρες. Στην Πορτογαλία αυτό συμβαίνει. Παραμένουν λίγες εβδομάδες και μετά τηλεφωνούν από τη Γερμανία γενικά για να μας ευχαριστήσουν ότι σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, ήσασταν υπέροχοι Πορτογάλοι, αλλά τώρα είμαστε στη Γερμανία γιατί εκεί θέλαμε να πάμε. Και χρησιμοποίησαν το μηχανισμό της μετεγκατάστασης για να φτάσουν στη χώρα που από την αρχή ήταν ο προορισμός τους. Άρα ο μηχανισμός αυτός ακόμα έχει ε, πολλές ατέλειες και προβλήματα για να μην μιλήσω για τη βραδία εφαρμογή. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ακούσαμε ότι πολλά από τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Ενώ μπορεί να έχουμε μεσολαβήσει χρόνια ολόκληρα ε, με παραμονή τους στο Λίβανο, στη Συρία, ε, στην Ιορδανία μάλλον, στην Τουρκία. Και έρχομαι τώρα στην ερώτησή μου. Τι γίνεται με την κοινότητα των Γεζιντή που ήταν και θύμα γενοκτονίας. Υπάρχει ειδική μεταχείριση για τους γεζιντή. Αυτοί ήταν σε καταβλισμούς όπου άνδρες, γυναίκες, παιδιά είχαν ζήσει δράματα, είχαν τραύματα χωρίς καμία ε, ψυχολογική υποστήριξη για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα τραύματα αυτά. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου και οι ερωτήσει μου. Αναγνωρίζω βεβαίως ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, αλλά παραμένουν κάποια πολύ ανισχυτικά φαινόμενα. Και μιλώ για κάποιες λειτουργίες ε, ε, στην εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου και αυτό καθυστερεί τόσο πολύ και η οικογενειακή επανένωση. Και έτσι εξηγούνται και διάφορα άλλα προβλήματα που βλέπουμε σε όλη τη διαδικασία. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ορισμένε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εθελοντική επιστροφή. Ε, Επικουρούμενη φυσικά από, από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης έχουν δημιουργηθεί κάποια θέματα με αυτή την εθελοντική επιστροφή. Αναφέρομαι στην ε, επιστροφή της χώρας προέλευσης ενός Αιθίωπα του μετόπου Ρώμα ο οποίος ε, έξι μήνες μετά από τη Λέσβο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Άντις όπου υπέστη σκληρά βασανιστήρια ε, τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και ένας Ιρανός υποψήφιος για τη λεγόμενη εθελοντική επιστροφή. Κινδυνεύει και αυτός με το ίδιο φαινόμενο. Σχετικά τώρα με την μετεγκατάσταση. Νομίζω ότι γενικά, προσωπικά, δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξη γιατί βλέπω ότι φτάνουμε κοντά πια στο Σεπτέμβριο, λίγη η περίοδος και ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Το λέγω αυτό γιατί αυτό το οποίο θα με ενδιέφερε είναι να γνωρίζω το τι θα ακολουθήσει. Τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει, ένα νέο πρόγραμμα μετεγκατάστασης να περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το νέο Δουβλίνο που θα ακολουθηθεί από ένα νέο σύστημα. Θέλω να προσπαθήσω ε, να κατανοήσω ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα πιο δύσκολα σημεία τα οποία τελικά κατέστησαν αυτή τη διαδικασία τόσο προβληματική. Τώρα η οικογενειακή επανένωση για την Ελλάδα ε, δεν είναι... Εγώ χαίρομαι που ο κύριος Βεβέη, εν περιπτώσει εύχεται να υπάρχει μια πιο γρήγορη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, αλλά δεν είναι ένα τυχαίο πρόβλημα. Η οικογενειακή επανένωση πρέπει να, έχει κάθε, να τύχει κάθε προτεραιότητας. Εσείς γνωρίζετε κύριε Βέβελ ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στη γερμανική κυβέρνηση και την ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να επιβραδυνθούν με δραστικό τρόπο οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης με πρόσωπα που πρέπει να πάνε από την Ελλάδα στη Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με την γερμανική κυβέρνηση για να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε αυτή η πίεση από πλευρά της παραβιάζοντας τους κανόνες του Δουβλίνου και του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή. Ε, μία άλλη ερώτηση, πάντα για το θέμα της επανεγκατάστασης. αναφέρεται κυρίως στην Ιταλία ανάμεσα στις αντιρρήσεις οι οποίες προβάλλονται στα αιτήματα τα οποία κάνει η Ιταλία περιλαμβάνονται επιχειρήματα σχετικά με την δημόσια ασφάλεια. Υπάρχει δηλαδή μια ρήτρα η οποία χρησιμοποιείται στο, στη διαδικασία λήψης απόφασης. Οι αιτίε άρνησης, οι οποίες να βασίζονται στο επιχείρημα της δημόσιας ασφάλειας, δεν επεξηγούνται με βάση μια μεμονωμένη μελέτη του συγκεκριμένου προσώπου στο οποίο αρνείται η μετακίνηση αυτή. Οπότε κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν η διαδικασία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη ή πράγματι μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Είναι πολύ πιθανό. Εφόσον λοιπόν, ειδικά για την Ιταλία, υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας σε σχέση με την άρνηση, Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια επαλήθευση ανεξάρτητη των αιτίων τα οποία προκαλούν την συγκεκριμένη και οδηγούν στη συγκεκριμένη άρνηση. Πάντα για το ίδιο θέμα. Αυτός ο οποίος ζητά άσυλο, ο οποίος είναι υποψήφιος για μετεγκατάσταση, ε, δεν λαμβάνει ή λαμβάνει με πολύ μεγάλη χρονική στέρηση τα τεκμήρια, τα τμήματα εν πάση που συναποτελούν τον προσωπικό του φάκελο. Δεν είναι δηλαδή εν γνώση των στοιχείων και της τεκμηρίωσης ε, με βάση τις συνεντεύξεις που προηγήθησαν. Αυτή η έλλειψη εγγράφων είναι αυτό το οποίο πολλές φορές παρεμποδίζει την οικογενειακή επανένωση γιατί στις νέες χώρες δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει την οικογένειά του σε μια άλλη χώρα. Και τώρα έρχομαι στα της Τουρκίας. Και θέτω το ερώτημα στον Δ. Βερβέλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα από την ελληνική κυβέρνηση να τροποποιήσει τις νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ελλάδα έτσι ώστε να επιτραπεί η παλινόστηση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις των λεγόμενων ευάλωτων κατηγοριών. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο αίτημα. Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει ως έχει. Και μάλιστα όταν λέγεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίζει κανείς τα λεγόμενα ιδιαίτερα ευάλωτα πρόσωπα, είναι σαφές ότι η νέα διαδικασία προβλέπει ότι η έλεγχη αυτή θα πρέπει να γίνεται δύο με τρεις ημέρες αμέσως μετά την άφηξη των συγκεκριμένων αυτών προσφύγων ή μεταναστών. Όλα αυτά πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και αυτό το εξήγησαν ο και η Human Rights Watch και άλλες ΜΚΟ. Είναι αδύνατον σε δύο-τρεις μέρες να κάνει κανείς μια τέτοια πλήρη αξιολόγηση. Και μια τελευταία ερώτηση πάντα σχετική με την Τουρκία. Η δήλωση με την Τουρκία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή δήλωση αν θέλετε, στην Ελλάδα είναι υποψήφιοι για τη μετεγκατάσταση μόνο αυτοί οι οποίοι είναι παρόντες στην χώρα από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2015 μέχρι τις 15 Μαρτίου του 2016. Την ημέρα που υπεγράφει αν θέλετε αυτή η συμφωνία ή η δήλωση έστω με την Τουρκία. Σας υπενθυμίζω ότι έχει υπάρξει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο αμφισβητεί αυτή την χρονική περίοδο, την περιορισμένη χρονική περίοδο πέραν της οποίας δεν θα επιτρέπονται πλέον μετεγκαταστάσεις. Διαρωτώ με λοιπόν η Επιτροπή και η κυβέρνηση ελληνική πώς αντέδρασαν στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαρωτώ αυτή η απόφαση είναι νόμιμη το να σταματούν οι μετεγκαταστάσεις την 16η Μαρτίου του 2016. διότι η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας δεν είναι μια νομικά δεσμευτική αν θέλετε πράξη, το λέει η ίδια η Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Ζήπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ίσως με δύο μικρές ερωτήσεις που έθεσαν και κάποιοι συνάδελφοι. Ερώτηση πρώτη. Στην Ελλάδα ισχύει ότι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και άτομα που ανήκουν σε αυτές θα πρέπει να έχουν τη μεταχεία διαδικασία για το άσυλο και ενδεχομένως ε, να μεταφέρονται και στην υπηρετική Ελλάδα και όχι να παραμένουν στα νησιά. Και καλά κάνει και ισχύει αυτή η ε, νομοθεσία, αλλά φαίνεται ότι μετά από πίεση έχει αλλάξει. Επίσης, αν πάρεις απορριπτική απόφαση και θέλεις να κάνεις προσφυγή, μπορεί να χάσεις την ευκαιρία να υποφεληθείς από ένα υποβοηθούμενο ε, σύστημα εθελοντικής επιστροφής και ένταξης. Όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα που συμβαίνουν, μας οδηγούμε στο να αποκομίσουμε την εντύπωση ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά δεν είναι να βοηθήσουμε την Ελλάδα, ούτε να βοηθήσουμε τους μετανάστες, αλλά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι καλύτερα να μην φτάνετε καθόλου στην Ευρώπη, γιατί δεν σας στέλνουμε εδώ. Και θα προσθέσω και μια μικρή πολιτική δήλωση που δεν στρέφεται κατά των δύο ομιλητών μας σήμερα, αλλά Πραγματικά πιστεύω ότι είναι απίστευτο αυτό που κάνουμε με τη χώρα αυτή, το κράτος μέλος που λέγεται Ελλάδα και τους μετανάστες που θέλουν να βρουν μια νέα προοπτική. Ε, από το 2008 που είχαμε αυτή την οικονομική κρίση είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έπρεπε να κάνει ε, κάποια πράγματα αλλά ε, είναι υπό μεγάλη πίεση. Πρέπει να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Έμαθα αυτή τη βδομάδα ότι θα πρέπει και το νερό και το φυσικό αέριο, έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας, οι συντάξει έχουν περικοπεί πάρα πολλές φορές και η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί για πρώτη φορά να δημιουργήσει ένα στοιχειώδη σύστημα ασύλου και δεν τους βοηθάμε. Θέλουμε να κρατήσουν όλους αυτούς τους ετούντες άσυλο ή να τους επιστρέψουν στην Τουρκία. Ήρθε εδώ το Συμβούλιο και δεν είχε καμία λύση για τη μετεκατάσταση. Όλοι διαμαρτύρονται και οδύρονται ότι έχουμε γεμίσει μετανάστες. Μα πώς σας ήλο έχουμε στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Πολωνία, στη Σλοβενία. 20. Έχουν φτάσει στους 100 μήπως. Ζητώ συγγνώμη που τα ακούτε εσείς τώρα. Ξέρω ότι είστε νέο μέλο και νέα κράτη-μέλη και πρέπει να δείτε κι εσεί πώ θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Αλλά αυτά που ακούμε από το Συμβούλιο είναι απίστευτα πράγματα. Και ταυτόχρονα είδα και ένα μήνυμα από τον κύριο Βέμπερ, πρόεδρο μεγάλη πολιτική ομάδα εδώ, που μα λέει ότι η επιπλέον βοήθεια για την Ελλάδα θα πρέπει να δοθεί μόνο αν αλλάξει κυβέρνηση. Απίστευτα πράγματα. Και πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να στέλνουμε τέτοια μηνύματα ούτε να, να με τέτοιο τρόπο. Αλλά για τον κύριο Βέμπερ και τον κύριο Σόιμπλε και άλλους, ακόμα και ε, το ο, ο Διεθνής Οργανισμός ε, θεωρείται ε, το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το θεωρούν αριστερό, σοσιαλιστικό ίδρυμα. Δεν είναι τίποτα αριστεριστές αυτοί, ούτε ε, είναι φιλάνθρωποι. Αλλά λένε για το χρέος ότι θα πρέπει να περικοπεί γιατί δεν υπάρχει προ, ε, προοπτική εκτός από την ευελάφρυνση του χρέους. Και βγαίνουν αυτοί και λένε αλλάξτε κυβέρνηση. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσετε εσείς, διότι δεν έχετε και την άδεια να το κάνετε. Αλλά ποια μηνύματα στέλνουμε στα άλλα κράτη-μέλη και τους ετούντες άσυλο. Για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από τα βασανιστήρια, από τις διώξεις και έρχονται στην Ευρώπη και εμείς τους λέμε «Α, ζητούμε συγγνώμη, έχουμε πολλά προβλήματα δικά μας». Και να προσθέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένως να καταρτήσει ένα κατάλογο. Πόσα χρήματα έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για να χτίζουμε φράχτες, να προστατεύουμε τα σύνορά μας, δίνουμε λεφτά στην Τουρκία για τη συμφωνία με την Τουρκία, πόσα χρήματα διαθέτουμε στο Αφγανιστάν, επενδύουμε για την σύνοροφυλακή και την ακτοφυλακή και πόσοι μετανάστες θα μπορούσαν να είχαν βοηθηθεί από τα χρήματα αυτά για να ενταχθούν και για τις αιτήσει ασύλου τα επόμενα χρόνια. Και το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι Sorry, δεν έχουμε εμεί καμία ευθύνη. Φροντίστε εσείς εκείνους που ζητούν άσυλο. Και κάνουμε μια συμφωνία ε, όπου σπρώχνουμε την Ελλάδα σε μια ολέθρια κατάσταση και την αφήνουμε στη μοίρα της. Ξέρω ότι δεν φταίτε αλλά έπρεπε να τα πω πώς να τα εκπέμψω αυτά προς το Συμβούλιο. Για άλλη μια φορά, το Συμβούλιο δεν επέδειξε την προθυμία να βρει λύση, να αναλάβει τις ευθύνες του από κοινού, όχι μόνο για να αλλάξει η κατάσταση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του κακού της αναγκαστικής μετανάστευσης, αλλά και να επιμεριστούμε καλύτερα τις ευθύνες και το βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κρίμα για μένα αυτό και θέλω να δω μια πολύ διαφορετική ένωση και σε αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σταχόφσκι. Κυρία Σίπελ, μάλλον ονειρεύομαι. Με κοροϊδεύετε. Νομίζω ήταν πολύ διασκεδαστικά αυτά που μας είπατε. Επικρίνετε την τσεχική δημοκρατία, λέτε ότι η τσεχική δημοκρατία σταμάτησε να δέχεται πρόσφυγες. Ξέρετε ποιος το σταμάτησε, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση. Εσείς ποιανού συντονιστής είστε των σοσιαλιστών, κυρία Ζήπελ. Πότε θα έρθετε εσείς στην Τσεχική Δημοκρατία για να τα εξηγήσετε αυτά στον Πρωθυπουργό Σομπότκα και στον Υπουργό Εσωτερικών και να τους πείτε ότι τους επικρίνετε. Ε, παράσταση για μας εδώ στην αίθουσα είναι αυτή. Σας ε, παρακολουθούσα εγώ κυρία Σίπελ, μην βγάζετε τα ακουστικό σας. Ξέρω ότι δεν ε, καταλαβαίνετε τσεχικά και αν θέλετε να παίξουμε θέατρο εδώ, αντί να λύσουμε τα προβλήματα, τότε θα πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Οι σοσιαλιστές είναι αυτοί οι οποίοι σταμάτησαν την μετεγκατάσταση στην χώρα μας. Το, ε, το κόμμα μου, οι, σοσιαλδημοκ... οι ήθελαν να κάνουμε μετεγκατάσταση και ψάχναμε να βρούμε και κόσμο να τον βοηθήσουμε να μετεγκατασταθεί στη χώρα μας. Να σταματήσουμε τώρα τις πολιτικές φανφάρες και να δούμε λίγο και τα στοιχεία. Ναι, συνολικά έχουμε περίπου 20.000 άτομα τα οποία μετεγκαταστάθηκαν. Γιατί δεν έχουμε περισσότερους. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ε, καταγράφησαν ως άτομα προς μετεγκατάσταση στην ε, Ανατολική Ευρώπη από την Ελλάδα και την Ιταλία χάθηκαν. Γιατί δεν μπόρεσε κανείς να τους βρει. Και αυτή είναι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να μας δώσετε μια απάντηση και μάλιστα χωρίς συναισθηματισμούς. Και μία ακόμα ερώτηση από πλευρά μου. Η Λιθουανία και οι μετεγκαταστάσει εκεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι μετεγκαταστάθηκαν στη Λιθουανία έφυγαν για άλλη χώρα. Πώ έγινε αυτό, μάλιστα για τη Γερμανία πιο συγκεκριμένα, στην οποία πλέον διαμένουν μόνιμα. Πώ θα το επιλύσετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Και τώρα θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Μίλλερ ως επικεφαλής αντιπροσωπείας. Αν δεν θέλετε να προσθέσετε τίποτα στην έκθεση, όχι για την έκθεση, αλλά επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τη συζήτηση, διότι νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος όταν συζητάμε ποιο κόμμα τώρα εδώ ε, ήταν το πιο αποτυχημένο, οι χριστιανοδημοκράτες ή οι σοσιαλιστές, δεν είναι συζήτηση αυτή. Πρέπει να δούμε το θέμα ως ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι θέμα κομμάτων. Ε, αν απλώς λέμε ότι φταίει το ένα ή το άλλο κόμμα, δεν βρίσκουμε λύση. Εμείς εδώ λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση. Και νομίζω ότι το θέμα εδώ είναι σαφές όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και τα εθνικά συστήματα, ο τρόπος των κρατών μελών δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή λύση επί του θέματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτος ο κύριος Νίλσεν. Ναι, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τα σχόλια και τις ερωτήσεις θα προσπαθήσω να καλύψω τα θέματα της μετεγκατάστασης. Καταρχάς, όσον αφορά το πού βρισκόμαστε και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Και την ερώτηση της κυρίας Ένστ. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20.000 άτομα 10.000 άτομα συγγνώμη, στην Ελλάδα, τα οποία είναι προς μετεγκατάσταση. Ε, φέτος είμαστε περίπου 2 με 2.500 άτομα το μήνα ε, θέλουμε να φτάσουμε στους χονδρικά 3.000 ανθρώπους το μήνα και θα μπορέσουμε ίσως να έχουμε μετεγκατάσταση ε, για τα άτομα που είναι στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της ε, απόφασης μετεγκατάστασης. Να έχουμε βεβαίως κατά νου ότι οι υποχρεώσεις των κρατών μελών που αναφέρονται στην έκθεση δεν ολοκληρώνονται και δεν ακυρώνονται στο ε, τέλος Δεκεμβρίου του, 17, του Σεπτεμβρίου του 2017, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κάποιοι είπαν ότι τα πράγματα προχώρησαν πολύ αργά και δεν έγινε και αρκετά μεγάλη πρόοδο. Ε, δεν νομίζω ότι τώρα πρέπει να κάνουμε απολογισμό τη διετού εμπειρία. Η διαδικασία ξεκίνησε πολύ αργά και τα κράτη-μέλη άρχισαν να αναλάβουν τι δεσμεύσει του. Ε, Επομένω, ε, προχωρήσαμε πάρα πολύ αργά. Το τελευταίο τρίμηνο όμω κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι στόχου μπορούμε να πετύχουμε για να μετεγκατασταθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταγραμμένου καταλόγου προς μετεγκατάσταση. Τώρα, Κατά την άποψή μας, οι συνθήκες στην υπηρετική Ελλάδα για τα άτομα τα οποία είναι προς μετεγκατάσταση είναι ικανοποιητικέ, Υπάρχει χώρος για όλους και με τη βοήθεια της ΥΠΑ για τους πρόσφυγες. Ε, πολύ εύστοχη παρατήρηση ότι κάποια κράτη-μέλη φαίνεται να ε, εκμεταλλεύτηκαν ε, την ασφάλεια ως πρόσχημα για να απορρίψουν κάποιες αιτήσει. Ε, ε, τα είδαμε και αναλυτικά σε προηγούμενες εκθέσεις. Ενθαρρύναμε κάποια κράτη-μέλη και το κάνουν αυτοί κάποια κράτη-μέλη όταν ε, επικαλούνται την ασφάλεια θα πρέπει να δίνουν και λόγους. Για παράδειγμα η Ιταλία. Ε, για ποιο λόγο αρνείται τη μετεγκατάσταση κάποιου για λόγους ασφαλείας. Κάποια κράτη-μέλη δυστυχώς δεν ακολουθήσαν τη συστασία και δεν δίνουν αιτιολόγηση και αυτό φυσικά μας οδηγεί και σε υποψίες ότι χρησιμοποιείται ω πρόσχημα. Τώρα, μετά τις 26 Σεπτεμβρίου δεν θα μπορώ να σας πω εγώ τι θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν έχει σχέδια για παράταση των σχετικών αποφάσεων, αλλά νομίζω ότι η εμπειρία καταδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει ε, πρόοδος για την λεγόμενη πρόταση του Δουβλίνου, τη νέα πρόταση. Θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή ε, συνιστόσα ε, και να υπάρχει πρόταση από τους συνομοθέτες, διότι αυτό είναι το πιο απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Κάτι τελευταίο από πλευρά μου για την επανένωση των οικογενειών. Ε, έχουμε διαπιστώσει ότι και αυτέ οι διαδικασίε προχωρούν σχετικά αργά στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καταφέρει βάσει των πληροφοριών που έχουμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει άμεση παραβίαση ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από τα κράτη-μέλη, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ο αριθμό των υποθέσεων από ό,τι στο παρελθόν και αυτό φυσικά είναι πίεση για τι εθνικέ αρχέ και δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν τι υποθέσει. καποια Κάποια κράτη-μέλη, για παράδειγμα η Γερμανία, προσπάθησαν να ε, οργανώσουν το θέμα διμερώς ε, με την Ελλάδα για να, τον αριθμό των υποθέσεων που θα διεκπαιρεώνουν το μήνα και ε, μέσα σε πιο χρονικό διάστημα. Αυτό επιτρέπεται βάσει του Δουβλίνου 3 να αποφασίζουν δηλαδή διμερώς τα κράτη-μέλη και να συμφωνούν πώ θα γίνεται η διαδικασία. Ε, είναι όμως βραδία η διαδικασία, αλλά φαίνεται να λειτουργεί τουλάχιστον από νομική σκοπιά. Ε, εξακολουθούμε να τα παρακολουθούμε τα πράγματα, αλλά η συνολική αριθμή για την επανόνωση ε, οικογενειών είναι αρκετά υψηλή. Είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι μεταφέρθηκαν εκτός Ελλάδος βάσει αυτής της διαδικασίας. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω στα προηγούμενα σχόλια. Ποιος αποφασίζει για να υπάρξει κράτηση και ε, τι μέθοδος ακολουθείται. Εδώ είναι εθνική αρμοδιότητα, αυτό το κάνουν οι εθνικές αρχές οι οποίες αποφασίζουν πάνω σε αυτό, στα κέντρα κράτησης. Είπα ήδη ότι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε μια διαφορετική άποψη, αλλά θα θέλω να είμαι ειλικρινής και να εξηγήσω γιατί οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την πρακτική που ακολουθούν μέχρι τώρα. Η λογική της νομικής ρύθμισης είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιος ζητά να υπάρξει εθελοντική επιστροφή αποσύρει ταυτόχρονα την αίτησή του για την χορήγηση ασύλου. Οπότε από αυτή τη στιγμή και μετά δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραμείνει νόμιμα στην χώρα. Το λέω λίγο αν θέλετε χονδροειδώς, αλλά σε αυτή την περίπτωση οφείλουν οι ελληνικές αρχές να προχωρήσουν στην κράτηση του προσώπου άνδρα ή γυναίκας. Θα προτιμούσαμε όμως να βρεθεί μια διαφορετική μέθοδος και το συζητάμε άλλωστε αυτό με τις ελληνικές αρχές τώρα. Για την ε, εθελοντική ε, επιστροφή είναι σαφές. Ε, θα πρέπει να αποφασίσουν ή να ζητήσουν άσυλο ή να ζητήσουν εθελοντική επιστροφή ε, αυτό δεν είναι όμως αλήθεια ότι το έχουμε επιβάλει ένα από τα δύο. Πρέπει να είμαι σαφής αυτό. Το θέμα δεν είναι να γίνει μια επιλογή, αλλά πρακτικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αν ζητείς ε, να υπάρξει επανεξέταση της αίτησής σου για άσυλο, τότε χάνεις το δικαίωμα επιστροφής. Κοιτάξτε να σας εξηγήσω λίγο πώς έχει η κατάσταση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πρακτική. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η τεράστια πλειοψηφία των προσώπων αυτών ζητούν άσυλο πρώτα, σε μια πρώτη φάση και στη συνέχεια μπορούν να καταγραφούν και μετά το αίτημά τους αυτό για την εθελοντική επιστροφή. Αυτή τη στιγμή το κάνουν αυτό ε, θα πρέπει να αποσύρουν την πρώτη τους αίτηση για το άσυλο. Αυτή άλλωστε είναι η λογική. Αν κάποιος δεν μπορεί να παραμείνει στην Ελλάδα νόμιμα, δεν πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα. Υπήρξε επίσης και μία ερώτηση για το ποιος είναι τελικά υπεύθυνο. για την εφαρμογή του συστήματος επιστροφής στην Τουρκία. Αυτό το οποίο προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ότι τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να έχουν τέτοιου είδους προγράμματα εθελοντικής επιστροφής, αλλά δεν διευκρινίζουμε εμείς το πώς θα γίνει αυτό σε κάθε χώρα. Η ερώτησή σας λοιπόν για το ποιος αποφασίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ελληνικές αρχές. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες σύμφωνα με την πίεση που ασκεί η Επιτροπή προς τις ε, ελληνικές αρχές να στέλνει τις ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες ή ηλικιακές κατηγορίες στην Τουρκία. Κατανοώ το από πού προέρχεται αυτή η διαπίστωση. Να σας διευκρινίσω λοιπόν το πώς έχει πραγματικά η κατάσταση. Τμήμα του κοινού προγράμματος δράσης, το οποίο είχαμε συμφωνήσει με τον Υπουργό τον κύριο Μουζάλα, ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε αποφασίσει είναι ότι θα έπρεπε να εξεταστεί το εάν. Αυτό μπορεί να συμβεί δίδοντας τις απαραίτητες εγγυήσει εκεί όπου αυτό απαιτείται. Αυτό είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα δράσης. Αυτό διερευνήθηκε στη συνέχεια και οι ελληνικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για διάφορους λόγους δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιστροφή κάποιων ευάλωτων κατηγοριών, αλλά αυτό το οποίο αποκλείεται είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας επιταχυμένης διαδικασίας. Γιατί ειδικά για τις ευάλωτες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές ρήτρες προστασίας. Αυτό γίνεται λοιπόν, αυτή είναι η κατάληξη αυτής της ε, ε, επικοινωνίας και στην πρακτική οι κοινωνικές αυτές κατηγορίες παραπέμπονται στην χρήση της κανονικής διαδικασίας. Τώρα, οι ΜΚΟ έχουν παραπονεθεί ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανείχνευση των ευάλωτων χαρακτηριστικών τμήματων των προσώπων αυτών. Ας προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε εδώ κάτι, ότι είναι προς το συμφέρον των ε, ευάλωτων αυτών προσώπων τα ευάλωτα χαρακτηριστικά τους να ανοιχνεύονται το ταχύτερο δυνατόν. Διότι αυτή τη στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε είναι σαφής η διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Και αυτό το οποίο συμβαίνει ότι ακριβώς λόγω αυτών των ευάλωτων χαρακτηριστικών οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μετακινηθεί από τις νησιωτικές περιοχές στην υπηρετική χώρα. Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή είναι κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει και μάλιστα σχετικά έγκαιρα. Πάντως το σύστημα αυτό το οποίο κάτι το χαρακτηρίζει θα έλεγα είναι η επιφυλακτικότητα. Εμείς έχουμε ανεπίσημες επαφές και συζητήσεις με τις ΜΚΟ που εργάζονται στον τομέα αυτό. Δεν θα σας το πούν δημόσια αλλά θα παραδεχθούν τελικά το ποια είναι η πραγματικότητα δεν υπήρχαν ε, γιατροί του δημοσίου διαθέσιμοι. Ουσιαστικά οι ΜΚΟ είναι αυτές που έχουν αναλάβει τις ιατρικές υπηρεσίες για την ανείχνευση των ευάλωτων χαρακτηριστικών και αυτό το οποίο ε, στην ουσία χαρακτηρίζει τη διαδικασία αυτή είναι η επιφυλακτικότητα. Ασυνόδευτη ανήλικη. Πάρα πολύ σωστά Πολλοί από εσά εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Είναι κάτι το οποίο λέγεται εδώ συχνά, είναι πραγματικά δύσκολο θέμα να διαχειριστεί κανείς, όχι λόγω έλλειψης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, προσπάθειας ή οτιδήποτε άλλο. Σας έχω ήδη πει παλιότερα ότι εγώ έχω συζητήσει με ΜΚΙΟ και τους έχω πει κοιτάξτε σας δίδουμε τα, τα πετούμενα χρήματα, βοηθήστε μας να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και μας είπαν δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο προσωπικό με συγκεκριμένες γνώσεις και είναι μια πολύ σημαντική δυσκολία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση ως έχει τώρα, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε, έτσι ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ε, υπάρχει ημέρημνα για αυτούς με το σωστό τρόπο. Υπάρχει ένα θέμα με, το, ε, με την κυδαιμονία όπως γνωρίζετε, ε, όπως ακριβώς λέγει και η έκθεση. Μένει να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμα έτσι ώστε να βελτιωθεί το σύστημα κυδαιμόνευσης αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Ευτυχώς οι ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις που παίζουν κάποιον πιο ανεπίσημο ρόλο συνδράμουν. Ε, πάντως ε, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τώρα ήθελα να επαναλάβω και δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, αλλά κάθε φορά που ακούω κάποιον να λέει ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι παράνομη, κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω, ακόμα και υπό την ιδιότητά μου, που δεν είμαι πολιτικός. Τι λέει η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ουσιαστικά, ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο και η διεθνή νομοθεσία θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Και το εφαρμόζουμε αυτό. Κάθε πρόσφυγας ή μετανάστης που φτάνει στην Ευρώπη έχει δικαίωμα ε, σε ξεχωριστή εξέταση ε, της περίπτωσής τους με όλες ε, τις εγγυήσεις και τις δικονομικές πρόνοιες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί κανείς να έχει ανησυχίες και σωστά ε, και δικαιολογημένα για την ταχύτητα. Σας είπα που βρίσκονται τα πραγματικά προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν ακολουθούμε κανόνες και νομοθεσίες. Γιατί τις ακολουθούμε. θα σταματήσω εγώ και με στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε. Ευχαριστώ. πολύ κατατοπιστικές και λεπτομερείς οι απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Βερβέη. Δικός μου ρόλος τώρα είναι να ρωτήσω τους συναδέλφους. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια θα θεωρηθεί τελική η έκθεση, αν δεν λάβουμε σχόλιά σας μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Ό,τι σχόλια έχετε και παρατηρήσεις παρακαλώ να τα διαβάσετε στη γραμματεία και σας ευχαριστώ και τους δύο για τα σχόλιά σας, για την ενημέρωση και τελειώσαμε εδώ. Επόμενη συνεδρίαση στις 29 του μηνός, 9 με 12.30 το πρωί και 2 με 5.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Καλό σας απόγευμα.